Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, να σας ε, πούμε καταρχάς τι γίνεται σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ένα σημείο έχουμε μόνο να συζητήσουμε, την έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο τρίτος τριμερής διάλογος για την ε, μεταγκατάσταση της ε, έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων έγινε χτες, τη Δευτέρα, στις 9 Ιουλίου από κοινού με την ε, ε, ομάδα της ΕΚΟΝ για την, και συζητήθηκε και η κατάσταση της, ε, του οργανισμού του Ευρωπαϊκού. Εμείς ασχοληθήκαμε με τον Οργανισμό Φαρμάκων και η ΕΚΟΝ με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τραπεζών. Συζητήθηκε λοιπόν το κείμενο. Το Κοινοβούλιο επανέλαβε την απέτησή του για μια πολιτική δέσμευση από όλα τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται για την αναθεώρηση των διαδικασιών, για την επιλογή των εδρών των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών και Φορέων και ζήτησε την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις φάσεις της διαπραγμάτευσης. Η Προεδρία παρουσίασε την ε, ενημερωμένη εντολή από την ΚΟΡΕΠΕΡ ε, δίνοντας μια δήλωση του Συμβουλίου στην οποία πήντησε το Κοινοβούλιο με μια αντιπρόταση αναφέροντας ρητά την πιθανή αναθεώρηση της κοινή δήλωσης και την εφαρμογή της ε, συνήθους ε, νομικής διαδικασίας για την επιλογή της έδρας του, του οργανισμού. Υπήρξε μια συμβαστική πρόταση ε, που πάει πέραν βέβαια της εντολής του Συμβουλίου και οι αντιπροσωπείες αποφάσισαν μέσω της γραπτής διαδικασίας και μετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις να ολοκληρώσουν ε, την ε, διαδικασία αυτή της διαβούλευσης. Αυτά λοιπόν για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις και τώρα μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας. Ωραία. Λοιπόν, καταρχά, εφαρμογή των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου, πρόταση κανονισμού για τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση ε, σιότσου μονής απόσταξης στην αγορά της Ένωσης, το οποίο παράγεται σε άμβικα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία. Ο, μόνο όποιος το πίνει μπορεί να ψηφίσει. Απαρτία έχουμε. Λοιπόν, για να ψηφίσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Annie drank it. No? It's closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα, ψηφίζουμε την ε, γνωμοδότηση για το πολιετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξηφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών 1967-2006 και 2017-2107. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10. Υπέρ, κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται.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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την, ε, το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Τώρα, ψηφίζουμε την έκθεση πρωτοβουλίας για την εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εισηγητή ο κύριο Πότσου. Ξεκινούμε με την τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 2, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 38 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. And Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Όχι, 69 καταπίπτει, 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είδα όλα τα χέρια. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. And ε, εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε και το 72. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. It's Πέρας. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ, την 76, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τώρα, πάμε στην τροπολογία 80. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 82. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 6 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Άγκρι 3 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Άγκρι 15 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε την άγκρι 15 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Άρχιδη ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Άγκρι 14 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Με προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Έχει κάποιος αντίρρηση με την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την ε, προφορική τροπολογία της παραγράφου 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 103. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 105. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την Άγκρι 22. Πέρας πληροφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την Άγκρη 23, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 117, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 118, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 118. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγρι 35 υπέρ κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την Άγκρη 35. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 136. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 137. Υπέρ, Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 137. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και την 138 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Είναι πολύ κοντά τα αποτελέσματα σίγουρα. Έτσι γίνεται συνέχεια σήμερα. Εγκρίνεται λοιπόν. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε. 141. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 140 καταπίπτει, 139 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 143 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 144 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 10 υπέρ, κατά, αποχές Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την Άγκρι 10. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άγκρι 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την άγκρι 12 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Άγκρι 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω το ίδιο, αλλά να το ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο παραπάνω. Άγκρι 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πάλι με μία ψήφο διαφορά θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Όντως μία ψήφος διαφορά. Εγκρίνεται. Άγκρι 30 υπέρ κατά, αποχές. Ε, το ΕΛΚ δεν σας βλέπω. Υπέρ, έτσι. Για πάμε ξανά. Άγκρι 30 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 149 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 και άγκρι 31 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά απόχέ, εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά αποχέ, απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά απόχέ, εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά αποχέ, απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 18 υπέρ. Κατά αποχές Να το ελέγξουμε παρακαλώ, γιατί δεν είδα πολύ καλά. Νομίζω ότι θα περάσει, αλλά ναι, με μία ψήφο πάλι. Εγκρίνεται λοιπόν. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 182 υπέρ. Α, καταπίπτει. Σωστό. Οι διάφορες καταπίπτουν. Πάμε στην 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 219. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη καταπίπτει. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, όχι, δεν γίνεται. Ε, το ΕΛΚ να σηκώνει τα χέρια του παρακαλώ. Ε, συμβαστική 19 μην καθυστερείτε. Λοιπόν, εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Α, βλέπω διήστανται οι απόψεις. Εντάξει. Ε, μην κάθεστε μπροστά μπροστά τότε. Λοιπόν, εγκρίνεται η 19 η συμβαστική. 2-13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.15 υπέρ. Κατά αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Απίστευτο. 2.16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 216. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.22 υπέρ. Κατά. Η ECR είναι κατά. Απορρίπτεται λοιπόν με τα ε, ε, άγκρι 40. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι. Κυρία Γκροστέτ. Η συμβαστική 1. Να την ελέγξουμε βεβαίως. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 1. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 8 υπέρ Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 56. Πέρας. Εγκρίνεται. Όχι, αυτή καταπίπτει. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 15, υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 22. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 29 καταπίπτει. Τροπολογία 30 και 31 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές το ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τα 45. Πέρας. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Πολύ με δύσκολευετε σήμερα. Να, δεν διαλέγετε μία πλευρά. Λοιπόν, ελέγχουμε τη 48. Ε, στρατηγικές αλλαγές γίνονται εδώ στις ψηφοφορίες σήμερα. Οι ECR και οι ε, σοσιαλιστές με τους πράσινους και το ΕΛΚ. Ε, πέρας ψηφοφορίας. Well, we lost, Mr. Ε, χάσαμε λίγο το μέτρημα. Λοιπόν, εγκρίνεται 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Την 52 ηλεκτρονικά. Πέρας. Και απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 57. Ωραία. Την 57. Την 57. Τι θέλετε να το ξανακάνουμε. Οκ, okay, πάμε πάλι για την 57. Ελέγχουμε την 57. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας και εγκρίνεται. This uh, Mr. Και αυτή ήταν λοιπόν η έκθεση του κ. Πόκ. Πολύ, πολύ, πολύ αμφιλεγόμενη. Δεν ήταν μεγάλη η πλειοψηφία στο αποτέλεσμα. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα και στην Ολομέλεια. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία τώρα. It's an initiative report. Έκθεση της πρωτοβουλίας. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ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 167. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Πώς είπατε. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Το ΑΕΛΚ και οι σοσιαλδημοκράτες ήταν στην ίδια πλευρά. Άρα αυτό τα λέει από μόνο του. 167 τώρα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 195 υπέρ. Κατά. Απόχε απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Βεβαίω. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά έναρξη. και πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 2-12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 2-14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.34 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλετε να το ελέγξουμε. Για καλό και για κακό. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον απορρίπτεται. Ελέγχουμε όμως ηλεκτρονικά. It's closed. Πέρασε. Απορρίπτεται. 3,57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.72 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 340 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 343. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.58 στον το τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 400 υπέρ μαζί με την 89 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Υπέρ. Κατά. απόχε εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Αλληλεία παράγραφος 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλληλεία παράγραφος 1. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3 της Ελίας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 6 τη Επιτροπή Ελία υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 469 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για την 469 παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. Σημειμαστική 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε σε τελογικές σκέψεις. Τραπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Α, συγγνώμη καταπίπτει. Η 2 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ε, ομάδα Unblock 4, 5, 6, 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την ε, υπαριθμό 10. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ε, έπρεπε να το ελέγξουμε όμως. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ. Υπέρ ή κατά. Πάμε πάλι. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ελέγχουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 18. Ψηφίζουμε. Και πέρασε. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά άποχες έλεγχος. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία, 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 35 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Αλληλεία σε τη σκέψη F. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. λογική σκέψη G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, λογική σκέψη η H. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η Ι τώρα. Σε δύο τμήμα. Τα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης. Ηλεκτρονικά. And the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Πετύχατε πολλούς συμβασμούς για την έκθεση. Μία άλλη έκθεση πρωτοβουλίας ε, για, τις ε, εναλλακτικές, για τα εναλλακτικά καύσιμα στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ονομαδότηση προς την τραν. Ε, συμβαστική 1 υπέρ, 2 τώρα, συγγνώμη, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται σας ευχαριστώ το 19 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ, α, συγγνώμη καταπίπτει, ευχαριστώ για την υπόδειξη, 32 υπέρ, κατά, αποχές, η άλντε τάσεται κατά, α, όχι υπέρ, εγκρίνεται, 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά. Η Άλντε ψηφίζει κατά. Απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές Οι σοσιαλιστές στάσσονται υπέρ, ελέγχουμε, ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 68 ξεχωριστή ψηφοφορία, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 71 υπέρ, κατά, αποχές, το ECR πώς ψηφίζει, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 82 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά στο σχέδιο γνωμοδότησης πέρας και εγκρίνεται Τώρα ψηφίζουμε για μία γνωμοδότηση κανόνες και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με την εναρμονιστική νομοθεσία για τα προϊόντα. 58 υπέρ. Κατά αποχές. Τι κάνει το ΕΛΚ. Ξανά. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Τι κάνει, τι κάνουν οι φιλελεύθεροι. Άλτε εγκρίνεται. 67. Ας ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε 57 πρώτο το τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Θέλετε να ψηφίσετε. Έχετε διάθεση. Πώς το βλέπετε. Πέρασε. Τέσσερις δεν θέλουν να ψηφίσουν. Ωραία. Καλά. Εγκρίνεται. Αν, αν όμως είχα ψηφίσει όλοι, μπορεί να ήταν άλλη η 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, ελέγχουμε 76. και πέρας και εγκρίνεται. 77-78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 79 ψηφίσουμε αφού είχε εγκριθεί προηγούμενη. 79 και 80 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 81 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83, α όχι, όχι. 84 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 και 87 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 και 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά. Τι μου είπατε. Α, ήταν παρόμοια, ταυτόσιμη με την προηγούμενη, εντάξει. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Άρχεται ψηφοφορία, πέρας και εγκρίνεται. 11, 101 και 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. σύνδυαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνονται. 13 και 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 108 υπέρ. Κατά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 κατά. Ελέγχουμε την 113, γιατί δεν ξέρουμε τι κάνουν οι φιλελεύθεροι. Πέρας, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές. Τι κάνουν οι φιλελεύθεροι, ψηφίζουν κατά. Τότε απορρίπτεται 116 και 117 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτονται. 118 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε. Οι φιλελεύθεροι φταίνε. Πέρας. Και απορρίπτεται πράγματι. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Ελέγχουμε την 120. Πέρας και εγκρίνεται. 123 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές Ελέγχουμε. 18. Έλεγχος. Πέρας και εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 135-36 υπέρ, κατά τι κάνουν οι σοσιαλιστές υπέρ. Άρα εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά αποχές τι κάνουν οι φιλελεύθεροι. Εγκρίνεται. Ωραία. Ελέγχουμε. 139. Ελέγχουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται πράγματι. 140-141. Α, καταπίπτουν. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 3 και 143 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 144 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε, εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 149-150 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 151 με προφορική. Υπάρχει κάποιος που αντιτάσσεται στην προφορική. Ωραία, ψηφίζουμε τότε 151 με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. 154. The Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 163 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας και εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές. Τι κάνουν οι σοσιαλιστές, ελέγχουμε. Πέρας και εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές Ελέγχουμε την 166. Πέρας. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 169 υπέρ, κατά Αποχές. Τι κάνουν οι φιλελεύθεροι. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 169. Α, την ψηφίσαμε. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 170 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 172. Πέρας και εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 και 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 41 και 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 44 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Τι κάνουν οι φιλελεύθεροι, τάσσονται υπέρ, ωραία εγκρίνεται. δύο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ένα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δύο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 50 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 4. Α, ελέγχουμε. 56 ελέγχουμε λοιπόν. Πέρας. εγκρίνεται κατά μία ψήφο. Νόμιζα ότι είχαμε την ίδια πλειοψηφία. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το τελικό κείμενο ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Really? <laughs> Double check. Okay, so the last one. Τελευταία λοιπόν, η προστασία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τι αρνητικές επιπτώσει του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιά. Είναι ψήφισμα. Ψήφισμα για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τροπολογία 34. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το ψηφίζουμε αυτό. Το ψηφίζουμε. Λοιπόν, συνολικά θα ψηφίσουμε. Όχι. 33. Θα ψηφίσουμε την 33. Ποιος είναι υπέρ της 33. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Όχι. 38. Υπέρ, κα, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ή όχι. Για να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. And closed. Πέρας εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές το ECR τι κάνει υπέρ εγκρίνεται άρα θέλετε να το ελέγξουμε όχι προχωρούμε στο 54 ποιος είναι υπέρ Συγγνώμη κυρία Ζόμερ, ποιο θέλετε να ελέγξουμε, το 50. Ωραία. Το 50 λοιπόν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 50. The vote is And it is Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στο 54. Εντάξει. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55 και 56 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, δεν ξέρω. 66, λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, γιατί δεν ήταν σαφές. Και πέρας και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Αλλά δεν είδα τα χέρια σας να είναι τόσο πολλά, γι' αυτό αναρωτήθηκα. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Άλντε, τι κάνετε. εγκρίνεται 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 και 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω τι να σας πω. Να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. And it's closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 89. Closed. And it is adopted. Πέρας εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 103 ε, υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 105 υπέρ, κατά αποχές, ε, 1 και 5 συγγνώμη, 2 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 3 και 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελογικές σκέψεις. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά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 Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Και κλείνουν και οι ψηφοφορίες μας για σήμερα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Enjoy the lunch. Καλό μεσημέρι θα σας ευχηθώ γιατί ολοκληρώσαμε και θα τα ξαναπούμε στις 2.30 γιατί θα έχουμε παρούσα την Υπουργό για θέματα υγείας και περιβάλλοντος. Τα ξαναλέμε λοιπόν στις 2.30.